και δεσμεύεται με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω συνάδελφοι ότι μια αντιπροσωπεία της Μαλαισιανής Ομοσπονδίας είναι παρούσα στα επίσημα θεωρία. Θα ήθελα να ευχηθώ το καλωσόρισε σε αυτήν την αντιπροσωπεία που καθοδηγείται από τον πρόεδρο της Ιερουσίας της Μαλαισίας Φον Μέγκ. Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια της Μαλαισίας είναι τακτικές. Είναι μια ζωηρή κοινωνία η Μαλαισία, μια ζωηρή οικονομία επίσης και ιδιαίτερα δραστήρια στα πλαίσια του ΑΣΕΑΝ. Γι' αυτό ακριβώς είναι μεγάλη χαρά που καλωσορίζουμε τους μαλαισινούς φίλους. Ελπίζουμε η επίσκεψή σας να είναι καρποφόρα και ενδιαφέρουσα. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μπροκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εκπρόσωποι της Κομισιόν και του Συμβουλίου,